συνεδρίαση και έχω μία ανακοίνωση. Έχει απευθυνθεί ένα αίτημα άρχης ασυλίας του κυρίου Ρόμπερ Ιβασίσκεβιτς από το πολωνικό κράτος ε, σε σχέση με μία διοικητικού τύπου παράβαση. Αποστέλλεται λοιπόν το αίτημα στην Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων που είναι